the busiest <laughs> committee, and it Λοιπόν, κάνετε κάποια δουλειά, πολλή δουλειά στην Επιτροπή όταν είσαστε πλήρη ενεργά μέλη της Επιτροπής. Χωρίς συναισθηματισμούς, πρέπει να πω ότι ήταν προνόμιο να δω το έργο των μελών. Επί πέντε χρόνια συνάντησα φίλους και από τα άλλα κόμματα. Και καμιά φορά πηγαίνουν και στραβά τα πράγματα. Διότι έχουμε συναισθηματικά φορτισμένα θέματα. Θέματα ταυτότητας. Αλλά αυτό επειδή νοιάζεται ο κόσμος για τα θέματα. Και έτσι δημιουργείται μια άλλη διάσταση. Το είδαμε με τη Σοφή όταν έθεσε το ερώτημα στο τέλος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ έχω εκπαιδευτεί πολύ καλά να αντιμετωπίζω όλες τις καταστάσεις Έβλεπα το ε, Newsnight. Ε, ήταν, ε, την είδα στο Newsnight χτε και ήταν πολύ ήρεμη. Γατούλα ήταν στο, στην εκπομπή την αγαπημένη. Δεν ξέρω, εδώ δεν είσαι, Σοφή, αλλά ήσουν γατούλα εκεί. πραγματικό προνόμιο που εργάστηκα εδώ, το προσωπικό, ανήκει στο όλο πακέτο αυτό. Το ανώτερο προσωπικό ανήκει σε ομάδα. Πρέπει να πηγαίνει στο, στους διαλόγους, κάνει προσπάθειες, καμιά φορά εξαντλητική κατάσταση, δύσκολες συζητήσει, ε, επίμαχα ζητήματα. Μην φεύγετε στο μέσο των ομιλιών. Μην φεύγει στο μέσο της ομιλίας. Ευχαριστώ το προσωπικό, το ανώτερο προσωπικό, τα ανώτερα στελέχη. Ξέρετε τι θέλω να πω. Τους τελευταίους μήνες της θητείας ε, ήταν εντατικές οι προσπάθειες. Ε, τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ το δικό μου προσωπικό. Άνταμ, Μαρία, Σελήν. Έκαναν πολύ καλή δουλειά, εργάστηκαν σκληρά και το υπόλοιπο προσωπικό που μας βοηθά στη Λίμπε. Η Λίμπε βλέπετε είναι η επιτροπή αυτή όπου ε, όλοι λένε ε, όπου πηγαίνετε λένε α είσαι στην επιτροπή αυτή πάντα που πηγαίνω λέμε ότι είμαστε καλή επιτροπή. Γιατί όλοι εκπλήσονται όταν λέμε ότι ανήκουμε στη Λίμπε. Να ευχαριστήσω τον Αντουάν της γραμματείας. Δρέπεται λίγο, είναι ένας πολύ σεμνός άνθρωπος. ξέρετε, δεν είμαι πολύ Βρετανός όπως βλέπετε. Ε, είμαι πολύ συναισθηματικός στην έκφραση του λόγου μου. Ε, και Πάντα λοιπόν ε, βλέπουμε ότι ο Αντουάν εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κοινοβούλιο, η ομάδα ήταν υπέροχη. Είχαμε ακροάσεις, τριμερείς διαλόγους, 20 ώρες δουλειάς, κάποιος πρέπει να εργαστεί. Απίστευτο το έργο που έκαναν. Τον ευχαριστώ τον Αντουάν. Ο βράχος ήταν, ο βράχος μου. Και τέλος, να πω, είστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελέσατε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ήταν καθοριστική δουλειά σε το Κοινοβούλιο. Επίμαχα, δύσκολα θέματα που συζητήσαμε. Καμία φορά δεν αρέσει στον κόσμο αυτό που κάνουμε, αλλά είναι αποφασιστική σημασία. Και το ιστορικό του έργου μας μιλά από μόνο του. Ευχαριστώ τα μέλη. Μεγάλο προνόμιο να σας βλέπω να εργάζεστε. Ψηφιακό τομέα, μετανάστευση, ιδιωτικότητα, το κράτος δικαίου. Και στην επόμενη θητεία θα δείτε αν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η Επιτροπή Λίμπε θα δείτε πόσοι θα θέλουν να συμμετέχουν στην Επιτροπή Λίμπε. Εκεί γίνονται τα πράγματα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Ήταν τιμή για μένα. Εύχομαι σε όλους που θα επανέλθουν ό,τι καλύτερο και εκείνους που θα επανέλθουν επίσης ό,τι καλύτερο. Δεν θα πω τι θα κάνω εγώ. Ποιος ξέρει. Εγώ θα προσέχω τι λέει το Συμβούλιο, ο ΤΑΣΚ κλπ και άμα μου πούν θα σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για μια υπέροχη πενταετία. Όχι, έχουμε ψηφοφορία τώρα. Πάμε στην ψηφοφορία. Μία ψηφοφορία, δόξα τω Θεώ. Απλούστατη ψηφοφορία. Ο κύριος Κοράου, ε ο συνήθως απουσιάζει. Καλώς. Δεν το λέω έτσι. Ε, δεν είναι κάτι κακό, αλλά μας αρέσουν οι παραδόσεις. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει. Τέλος. Ε, εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Τελική ψηφοφορία της Επιτροπής μας μετά από 5 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Τέλος Μα και θα προεδρεύσει το επόμενο τμήματος της ε, συνεδριάσεως και εγώ θα επιστρέψω, σας το υπόσχομαι. Δεν προσπαθώ να ξεφύγω. Uh, Αδελφοί, μετά από αυτή την πολύ ωραία ομιλία, συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Θα θυμάστε ότι την 4η Ιουλίου το Κοινοβούλιο έκανε 8 ψηφίσματα μετά την έκθεση ΛΥΒΕ για τις συστάσεις ε, της Κομισιόν για την επαναδιαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών για την ανταλλαγή δεδομένων με Europol και Ισραήλ, Αίγυπτο, Αργενία, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, Τινησία και Τουρκία για σκοπούς επιβολής του νόμου προφανώς και βεβαίως ε, ε, εισηγητής ήταν ο πρόεδρος για τις 8 αυτές εκθέσεις το Κοινοβούλιο υπέβαλε πολλές ε, συστάσεις και τόνισε ότι η συνένεσή του θα ήταν υπό τον όρο της ικανοποιητικής ε, εμπλοκής του σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 218. Εν τω μεταξύ το Συμβούλιο ενέκρινε και τις τελικές ε, διαπραγματευτικές οδηγίες η Κομισιόν. Ήδη ξεκίνησε διαπραγματεύσει με μια χώρα, την Τουρκία, και η διαπραγματευτική ομάδα της ε, Κομισιόν ήταν στην Άγκυρα αρχές της εβδομάδας ε, πέρα από αυτό και την σχετική ενημέρωση. Σημαντικό είναι να ενημερωθούμε για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και με τις άλλες 8 χώρες ε, για όλα αυτά. Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Σεσίλια Γουέπκλειτς, ε, επικεφαλής της Μονάδας για την Ανταλλαγή Αστυνομικών Πληροφοριών ε, για 10 περίπου λεπτά. Μετά θα δώσω τον λόγο στους και οδησηγητές και όποιον βουλευτή ενδιαφέρεται. Κυρία Λιγκλέτζ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων με την Τουρκία έλαβε χώρα αυτήν την εβδομάδα στις 9 Απριλίου. Οι συνάδελφοι ε, είχαν έναν πλήρη γύρο διαπραγματεύσεων το πρωί και χρησιμοποίησαν το απόγευμα για να επισκεφτούν την τουρκική αρχαία προσωπικό, προσωπικών δεδομένων. στις άλλες ε, στα χώρες. Ε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα διαπραγματεύσεις, οπότε δεν μπορώ να σας πω για το τι έγινε και δεν έγινε ακόμα. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να σας ενδιαφέρει είναι ότι τον Δεκέμβριο συναντηθήκαμε όλες αυτές τις χώρες και παρουσιάσαμε τις βασικές ιδέες και τον σκοπό των μελλοντικών συμφωνιών και τα βασικά ζητήματα που ήθελε να αντιμετωπίσει η Κομισιόν. Οπότε μπορώ να σύντομη όσον αφορά τις άλλες χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν είμαι σίγουρη εάν άκουσα κάποια ακριβή πληροφορία για τις ε, διαπραγματεύσεις. Γιατί καλό θα ήταν να γνωρίζουμε εάν τουλάχιστον έχετε κάποιο χρονικό πλαίσιο για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων και κατά την απόψή σας ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία της συζήτησης. Ίσως να μην άκουσα προσεκτικά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή και τα ποια είναι τα πιο δύσκολα σημεία στις ε, διαπραγματεύσεις αυτές, γνωρίζοντας βεβαίως πως η κατάσταση με όλες αυτές τις χώρες ε, είναι ε, διαφορετική για την καθεμία, αλλά δύσκολη. Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικό. Ε, κύριε Πρόεδρε, να επεκταθώ λίγο για αυτό το οποίο είπατε το τελευταίο. Σωστά είπατε ότι είναι διαφορετικές αυτές οι χώρες μεταξύ τους. Οπότε όσον αφορά τα πιο δύσκολα σημεία, αυτό εξαρτάται από την κάθε χώρα. Όπως ξέρετε, στο Ισραήλ είχαμε εκλογές Γι' αυτό το Ισραήλ δεν ήθελε να μπει σε διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο, δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εξαρτάται πολύ και από τις εσωτερικές ε, διαβουλεύσεις ε, της κάθε χώρας, όπου έχουμε ελάχιστη επιρροή. Προσπαθούμε να συμφωνήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά μέχρι στιγμής ε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά... Βεβαίω, το να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα θα μας διευκόλυνε, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, εξαρτάται και από τους συνομιλητές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Βλέπω ότι ο κύριος Τερικάμπρας είναι στην αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε ερωτήσει γιατί είστε ο ή Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, έχω... Έχω δέκα ερωτήσεις. Πρώτον, οι μηχανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και η ΜΚΟ έχουν επισημάνει τις τεράστιες ελλείψεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις περισσότερες, ε, αν όχι όλες τις χώρες αυτές, όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιωτικότητας επιπλέον. Οι χώρες αυτές δεν έχουν κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό υπάρχει πραγματικός κινδυνός τέτοιες συμφωνίες να ενισχύσουν την καταστολή στα καθεστώτα αυτά απέναντι στους ε, αντιφρονούντες. Ειδικά η Αίγυπτος ε, και το Μαρόκο είναι, και η Τουρκία είναι πολύ ανησυχητικές περιπτώσεις. Οπότε θα πρέπει οι οχτώ χώρες να συμμορφωθούν πλήρως με τις προδιαγραφές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στον νόμο και στην πράξη. Πώς θα διασφαλίσει η Κομισιόν πώς ε, θα πληρούνται αυτοί οι όροι. Και αν μου επιτρέπετε και άλλη μια ερώτηση. Καθώς πολλές από αυτές τις χώρες, όπως η Αίγυπτος, χρησιμοποιούν ε, τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας για να καταστήλουν ειρηνικούς πολιτικούς αντιπάλους και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς θα διασφαλίσετε ότι ο διαμοιρασμός και η μεταφορά δεδομένων από την Europol δεν θα διευκολύνει τις κατασταλτικές αυτές πολιτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να θέλει τον λόγο, οπότε έχει η κυρία Λίγκλετς τη δυνατότητα να απαντήσει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για αυτή την πολύ σημαντική ερώτηση θα ήθελα να υπενθυμίσω την εντολή του Συμβουλίου και τις διαπραγματευτικές οδηγίες μας που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά. Όσον αφορά τους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Με την Τουρκία, παραδείγματος χάρη. όπου συζητάμε και τη μεταρρύθμιση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητο για εμάς και για άλλες συμφωνίες που θέλουν να συνάψουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι ανησυχίες σας νομίζω ότι κατοπτρίζονται στην εντολή που έχουμε λάβει και τις συστάσεις ε, του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν αναπόσπαστο τμήμα της εντολής μας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό και να φροντίσουμε να αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Τερικάμπρας ίσως να μην είναι πολύ ικανοποιημένος με την απάντηση. Να προσθέσω κάτι. Σύντομη ερώτηση. Η Διεθνή Συμφωνία θα περιέχει όλες τις συστάσεις του υποπτικού φορέα την προστασία των δεδομένων και τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα συμπεριλαμβάνει η Διεθνή Συμφωνία. Απάντηση. Δύσκολη ερώτηση. Λέει η πρόεδρο, μάλλον. Δεν ξέρουμε από την αρχή ποιο είναι το αποτέλεσμα των διαργασιών, αλλά αν μπορείτε να απαντήσετε, πρέπει να ευθυγραμμιστώ με την ανάλυση της Προέδρου. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα. Προσπάθεια είναι όμως. Αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όπως είπα, αυτά είναι τα εργαλεία, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές. Ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία μόλις τώρα. και εντάσσονται οι συνομιλίες αυτές στην εντολή μας. Τώρα, σε ποιο βαθμό μπορεί να εξασφαλίσει κανείς ότι όλες οι συστάσεις θα καλυφθούν είναι και θέμα ερμηνείας και αξιολόγησης. Είναι κάτι που μαζί θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό πιστεύω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως να επενθυμίσω σε όλους και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα του Κοινοβουλίου να ενημερώνεται και να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας βάσει του άρθρου 218. Οπότε προσβλέπουμε σε περαιτέρω παράληψη πληροφοριών, παραλαβή πληροφοριών, συγγνώμη, οπότε καταφθάσουν είτε γραπτό την επόμενη εβδομάδα, τι επόμενε εβδομάδε, αν συμβεί κάτι, και ακόμα περισσότερο στην επόμενη θητεία όταν θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να είναι σαφές όμως. Ευχαριστώ για την πρώτη αυτή γενική εικόνα. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι μια παρουσίαση περί της ομάδας εργασίας της ΛΥΜΠΕ για τον έλεγχο του χώρου Σέγγεν. Προβλέπεται για τις 10 και το θέμα. Ο συνάδελφος ο κ. Κοέλιο που θα ασχοληθεί με την έκθεση δεν μπορεί να έρθει πριν από αυτό. Οπότε μικρό διάλειμμα μέχρι τις 11 παρα 20 πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ. So Um, Συνάδελφοι, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Είχαμε μια πολύ ωραία ομιλία του Προέδρου μας, του Κλοντ Μοράις, για την τελευταία συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ πριν αποχωρήσουμε για την προεκλογική εκστρατεία. Συμβαίνουν όμως ενδιαφέροντα πράγματα. Να καλωσορίσω τον νέο συνάδελφο, Κάνσο μετά τον Εβάντι Παντά που πήγε στο Εθνικό Κοινοβούλιο, τον διαδέχεται. Θα έχει κάποιες όμορφες τελευταίες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο και ίσως και κάποιες εβδομάδες μετά τις εκλογές. Θα δεις πώς εργαζόμαστε. Καλώς ήρθες στην Επιτροπή Λίμπε για αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο του του Λεχθέντος. Πάμε αμέσως στο επόμενο σημείο αφορά την ομάδα εργασίας για τον έλεγχο του Σέγγεν, των θεμάτων Σέγγεν. Μετά τη δημιουργία της ομάδας αυτής της εργασίας το 2016, υπό την προεδρία του Κάλλος Κοέλιο, η ομάδα υπήρξε πολύ δραστηρία, εξέτασε πολύ άριθμα έγγραφα που παραλαμβάνει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων Σέγγεν και συναφών ζητημάτων. Ο κύριος Κοέλιο μαζί με άλλους είχε πολλή δουλειά για το συγκεκριμένο σημείο. Αμέσως να δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο για να μας ενημερώσει για τις πρόσφατες εργασίες που έλαβαν χώρα. Κύριος Κοέλιο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με τα χαρά να σας ενημερώσω για τις εργασίες ε, της ομάδας εργασίας για τον έλεγχο του Σέγγεν. Όταν φτάνουμε στο τέλος της θητείας ε, ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Αυτή η ομάδα λοιπόν, η ειδική ομάδα, συνεδρίαζε σχεδόν κάθε μήνα. Ενημερωνόμασταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του Συμβουλίου και των κρατών μελών. Καλωσορίσαμε εκπροσώπους και διευθυντές της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και τις ομάδες για την έλεγχο των συνόρων, της Europol και της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενέκρινε και την πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση Σέγγεν το Κοινοβούλιο. Κατόπιν αιτήματος της ομάδας εργασίας έγινε αυτό και έχω την τιμή που είμαι εισηγητής σας. Σημαντική συνιστόσα των εργασιών είναι τα μέλη της ομάδας εργασίας και η γραμματεία. Πραγματικά είμαστε μια καλή ομάδα και ευχαριστώ γι' αυτό. Επιτρέψτε με όμως να εστιαστώ επί τριών σημείων που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας. Καταρχάς η ομάδα εργασίας ε, απέδειξε ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν για να υπάρχει η σωστή προστασία του μεγαλύτερου επιτεύγματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δηλαδή ελεύθερη μετακίνηση. Σε καιρού με προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σέγγεν, τώρα περισσότερο ποτέ η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι απαραίτητη. Όμως, το Κοινοβούλιο ήταν και παραμένει συχνά αντιμέτωπο με τα όρια του δυνατού όσον αφορά τις πληροφορίες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί μας παρέχοντας πρόσβαση. Όμως δεν είχαμε πάντα αυτό που επιθυμούσαμε, όσα επιθυμούσαμε, αλλά η συνεργασία ήταν καλή. Όμως η πρόσβασή μας στις πληροφορίες εξαρτάται κατά πολύ από τη δυνατότητα που έχουμε να επεξεργαζόμαστε ε, τις ομάδες των στοιχείων. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπινους πόρους γι' αυτό και καλύτερα εργαλεία για να γίνει σωστή αξιολόγηση και να δούμε πώς εφαρμόζουν τα συμπεράσματα τα κάτι μελη Δεύτερον, μετά τη δημιουργία της ομάδας εργασίας αυτής, ένα νέο μέσο δημιουργήθηκε, ε, η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα σύνορα, τα χερσαία και την ακτοφυλακή. Αντιμετωπίζουμε τεράστιο όγκλο πληροφοριών και χρειάζονται περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας για την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό το καινούριο μέσο συμπληρώνει το μηχανισμό ο Σέγγεν και είναι σημαντικό να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό σωστά. Τέλος, είμαι περήφανος για το έργο που επετέλεσε η ομάδα εργασίας είναι σαφές ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε συνέχεια στις δραστηριότητες αυτής της ομάδας την επόμενη θητεία. Το Κοινοβούλιο θα στείλει έτσι ισχυρό μήνυμα ότι το ρόλο μας για την προστασία του Σέγγεν τον παίρνουμε στα σοβαρά. Για αυτό το σκοπό λοιπόν τις επόμενες ημέρες προτίθεμε να συντάξω επιστολή προς τον πρόεδρο τον κύριο Μωράης παραθέτοντας τις δραστηριότητές μας και καθώς και το τι πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το μέλλον της ομάδας εργασίας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να ηγηθεί τη ομάδα η κυρία Βερζιά να συνεχίσει τις εργασίες να συνεχιστούν οι εργασίες τη ομάδα στην επόμενη θητεία, να συνεχίσουν προσπάθειε που έγιναν ε, για το Σέγγεν και χρειάζεται πολλά να γίνουν ακόμα. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε και τη συνεργασία. Thank you, Mr. for this. Ευχαριστώ κύριε Κοέλιο για την επισκόπηση των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε όσον αφορά τον χώρο του Σέγγεν. Έχω δύο συναδέλφους που θα ήθελα να μιλήσουν. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφο ε, Λόπες Αγγιλάρα. Ευχαριστώ Μπέργκερ και ευχαριστώ Κάρλος που κρατάς ζωντανή μέχρι την τελευταία στιγμή την Επιτροπή Λίμπε. Βλέπεις δεν είμαστε πολύ άριθμοι εδώ παρόντες, αλλά συνεχίζουμε. Και για να τα μίληψω ακριβώς την παρουσία σας εδώ, να μην περάσει έτσι ε, στα ψηλά, πράγματι, το είπατε πολύ σωστά, το Σέγγεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ευρωπαϊκής διαδικασίας που είχαμε ποτέ, αυτό που εκτιμούν ιδιαίτερα οι πολίτες και έχουν δίκιο. Σημαίνει πολλά η ελεύθερη διακίνηση και εξωτερικά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μόνη μου παρατήρηση είναι ότι έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να παραμείνει ζωντανό το Σέγγεν, το κεκτημένο αυτό του Σέγγεν. Εμείς, όχι το Συμβούλιο. Το Σέγγεν διεκόπη από διάφορες χώρες μέλη και το βλέπουμε κάθε φορά που πάμε στο Στρασβούργο, που είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν πάμε αεροπλάνο δηλαδή στο Στρασβούργο, μα ζητούν να δείχνουμε τα διαβατήριά μας ή τι ταυτότητές μας. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά. Εμείς κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Εγκρίναμε και το πακέτο διαλειτουργικότητα. το οποίο σημαίνει ότι το VIS, το SIS, δεύτερη γενιά, το ΕΚΙ, στο ΕΤΙΑ, στο Eurodac. Ακόμα και η ανταλλαγή φακέλων εγκληματιών είναι πράγματα που έχουν διασφαλιστεί μέσω της τεχνολογίας, μέσω των συστημάτων πληροφοριών τελευταίας γενιάς. Και αυτό για να μπορεί το Συμβούλιο να κάνει τη δουλειά του. Και τι είναι αυτό? Να επανέλθει το Σέγγεν παντού. Ελπίζω στην επόμενη θητεία και όσοι είμαστε εδώ και παραμείνουμε στη Λίμπε και όσοι νέοι έρθουν θα δείξουν ε, τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και εσύ Κάρλος προκειμένου το Σέγγεν να ξαναβρει ε, την ε, φόρμα του. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τα ευρωπαϊκά σύνορα, για την ακτοφυλακή. Πολλά συζητιούνται για τη Frontex που είναι βέβαια ξεπερασμένη. Τώρα υπάρχει μια νέα υπηρεσία. Πολλά λοιπόν ε, μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση και το Σέγγεν να ξανασταθεί στα πόδια του. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι και εγώ, σε αυτό το τελευταίο στάδιο εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αναγνωρίσω την ε, ποιότητα με την οποία δουλέψαμε υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών και να πω ευχαριστούμε. Για όλους εμάς πιστεύω ότι είναι τιμή που συμμετείχαμε σε αυτή την τόσο όμορφη περιπέτεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη υπέρ των αξιών που υποστηρίζει η Επιτροπή μας αυτή και όλα τη τα μέλη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Χουάν. Επόμενος η Μαρή Κριστίν Βερζιά. Παρακαλώ, Μαρή Κριστίν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι υποψήφια ξανά, οπότε είμαι σίγουρη ότι δεν θα είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία. Είναι επιλογή δικιά μου, καθαρά αυτή. Θέλω όμως να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους και το προσωπικό και τους διερμηνείς και όλους τους συνεργάτες μας από όλες τις πολιτικές ομάδες γιατί συνεργάστηκα με όλους τους και τους ευχαριστώ πολύ. Επί της ουσίας θέλω να ευχαριστήσουμε όλοι τον κύριο Κοέγιο. Το γνωρίζει ότι με ιδιαίτερη χαρά συνεργάστηκα μαζί του παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές έχουμε. Νομίζω ότι θέλουμε το χώρο Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία τόσο εκείνος όσο και εγώ. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε σε αυτή την ομάδα εργασίας προκειμένου οι χώρες να ξαναβρούν τη λογική τους. Και βεβαίως ευχαρίστως να συνυπογράψω την επιστολή αυτή μαζί του. Γιατί εγώ ζήτησα να αφήσουμε κάποια ίχνη από τη δουλειά που έχει κάνει η ομάδα αυτή εργασία σε αυτή τη θητεία. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους επόμενους, για την επόμενη θητεία. Το αποτέλεσμα του Σέγγεν απορρέει από την άρνηση του Συμβουλίου να διαπραγματευτεί πάνω στην έκθεση φαγιών. Και είναι κρίμα, γιατί είχαμε μια έκθεση απόλυτα λογική. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε τις χώρες να επαναφέρνουν εσωτερικά σύνορα όποτε θέλουν και για τους λόγους που θέλουν, Δυστυχώς αυτό γίνεται όμως από πολλές χώρες, χωρίς να υπάρχει κανένας τρόπος να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση, ενώ είναι ένα από τα βασικά κεκτημένα για τους Ευρωπαίους πολίτες στο Σέγγεν και έτσι νιώθουν την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στο χώρο Σέγγεν. Θέλω να πω στον κύριο Αγγιλάρ ότι αντίθετα με αυτόν εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε έχουμε καταφέρει το καλύτερο. Όχι, εγώ φοβάμαι ότι πάμε προς το χειρότερο και σας δίνω ραντεβού όσον αφορά τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων μετά από μερικά χρόνια. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι εδώ ε, ετοιμάζουμε μια βραδιφλεγή βόμβα. Μακάρι να αποδειχτεί ότι έχω λάθος. Αλλά αυτό μου λέμε είναι η λογική μου. Και νομίζω ότι έχουμε ετοιμάσει εδώ κάτι ε, του οποίου τις συνέπειες δεν είμαστε σε θέση ακόμα να εκτιμήσουμε και δεν καθίσαμε να ακούσουμε τις προειδοποίησεις από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από τις διάφορες υπηρεσίες ε, προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, επόπτη θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ. Τέλος κύριε Γκυλάρ, να σας υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχουν δύο έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει μία που είναι το Στρασβούργο, το προβλέπουν οι συνθήκε και αυτό δεν έχει αλλάξει. Αν εσείς θέλετε κάτι άλλο, τι να κάνουμε. Μπορεί να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, αλλά προς το παρόν η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι στο Στρασβούργο. Ακόμα και αν αυτό δεν σας αρέσει. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κυρία Πρόεδρε, Αντουάν, Κατρίν και σε όλους τους υπόλοιπους. Έτσι καλώς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα και ίσως και κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Παρόλο που αυτό δεν είναι το σημείο για συζήτηση για την μοναδική έδρα του Ευρωκοινοβουλίου, να επενθυμίσω τη σπάση ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αν έχουμε μία έδρα και αν μπορούμε να έχουμε μία έδρα και αν αυτή η έδρα που θα πρέπει να εδρεύει. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαστε εργαζόμενο κοινοβούλιο και δεν είναι θέμα πού είναι η έδρα του κοινοβουλίου, αλλά είναι τα άλλα θεσμικά όργανα με τα οποία μας συνεργαστούμε και πώς πρέπει να οργανωθεί αυτό. Μιλάμε λοιπόν για το χώρο Σέγγεν, έχοντας υπόψη αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Χουάν και Μαρή Κριστίν. Ίσως ο συνάδελφος Κάρλος Κοέλιο θέλει να επανακάμψει πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά, τον Χουάν Φερνάντο και τη Μαρή Κριστίν. Νομίζω ότι και οι δύο είπαν κάτι σωστό το πρόβλημα με την Σέγγεν δεν ήταν, δεν ήμασταν εμείς όπως είπε ο Χουάν Φερναντό εμείς στηρίξαμε τη Σέγγεν το Συμβούλιο ήταν και το Συμβούλιο υποστήριξε το, τη Σέγγεν όπως το κάνουμε εμείς ε, για την διαλειτουργικότητα είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ε, έκανε αυτό που μας ζήτησε η Κομισιόν τα ξέχασε το Συμβούλιο. Μιλάμε για έναν τομέα με τρεις διαστάσεις. Ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Και το Συμβούλιο κοιτάει μόνο την ασφάλεια. Η ελευθερία και η δικαιοσύνη δεν τους απασχόλησε πολύ. Και Χουάν Φερνάντο έδωσε ένα καλό παράδειγμα. Η νέα Frontex, η νέα υπηρεσία που πρότεινε η Κομισιόν. Και εμείς ευχαριστώς εγκρίναμε και ενέκρινε και το Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο με την υπηρεσία ασύλου. Γιατί δεν αφορούσε την ασφάλεια. Δεν υπήρχε η ίδια πολιτική πίεση. Και έχουμε κολλήσει. Χωρίς λύση. Κάπου μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και είναι κρίμα το ότι δεν είχαμε αποτελέσματα. Οπότε, όταν μιλάμε για τη Σέγγεν, μιλάμε για τον πυρήνα των αξιών μας και είναι μια μάχη που πρέπει ε, να δώσουμε με τον σωστό τρόπο και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι θα κάνουν σωστά την δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέλφους γιατί ε, γίνεται πολύ σκληρή δουλειά, έχουμε πολύ συχνά συνεδριάσεις και συχνά το κοινό δεν τα προσέχει αυτά. Ε, είναι όμως σημαντική δουλειά, θα είναι σημαντική γιατί όλοι συμφωνούμε ότι η ελευθερία μετακίνησης εντός της ζώνης Σέγγεν είναι ένα μεγάλο επίδεγμα που έχουμε και θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να συνεχίσει και στους τομείς ε, της ασφάλειας. Ε, ε, βεβαίως, αν δεν είχαμε ανοιχτά σύνορα εντός της Ένωσης, θα είχαν πολλές αρνητικές συνέπειες. Οπότε πρέπει να συνεχιστεί αυτό και ίσως στην επόμενη εντολή θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί εντός του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι το θεσμικό όργανο που είναι αδιαφανές πρέπει να δούμε και τον κανονισμό τους, γιατί δηλαδή ε, κολλάνε τόσο συχνά και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε τις δυνάμεις των κρατών μελών, τις εξουσίες τους, γιατί είναι τα μόνα οι μόνοι μπορούν να δρουν χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση που ίσως είναι πρόβλημα. Οπότε έχουμε περισσότερα μπροστά μας ε, εντός ε, της ζώνης Σέγγεν αλλά βεβαίως ε, και εντός των θεσμικών οργάνων. Οπότε θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ομάδα εργασίας. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα και για τους συναδέλφους ίσως που δεν θα επανέλθουν αλλά θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα πράγματα αυτά ακόμα και από μακριά. Πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Τώρα για δεύτερη φορά σήμερα έχουμε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου αναμένουμε ακόμα τους εισηγητές. Οπότε, ξέρω, κάντε καμιά βόλτα.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 So, dear colleagues, um, if you're ready, we can begin on point nine. Thank you to Mrs. Περνάμε στο σημείο 9, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για τις κοινοτικέ στατιστικές στην μετανάστευση. Η Σόφη αντικαθιστά εδώ την κυρία Βίλστρομ και σε ευχαριστώ Σόφη γι' αυτό. Η Σόφη λοιπόν θα μας ενημερώσει για την κατάσταση πραγμάτων των διοργανικών διαπραγματεύσεων στο φάκελο αυτό. Εγώ προείδρευσα στο τέλος και όντως είναι ιδιαίτερα θετική η εμπειρία μου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συμμετέχοντες. 31 Ιανουαρίου τον τελευταίο ο τριμερής διάλογος υπήρξε συμφωνία, αναβλήθηκε κάπως στην Κορεπέρε το Φεβρουάριο η έγκριση της συμφωνίας. Δημιουργήθηκαν προσδοκίες για έγκριση από πλευράς του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τώρα. Οπότε και πες μας, Σόφη, πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ, Κλόρτ. Θα διαβάσω τη δήλωση που μου έδωσε η Σεσίλια Βίλκστρομ που ζητά συγγνώμη που δεν είναι μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστεί τους και όδες εισηγητές και τους συνεργάτες τους για την εξαιρετική δουλειά που έγινε και που στήριξαν ε, το έργο στο φάκελο αυτό. Το, ο τελευταίος τριμές διάλογος, όπως είπες, έγινε στις 31 Ιανουαρίου και πετέχθη συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο πάνω σε ένα κείμενο. Στη συνέχεια πήγε το κείμενο στην Κορεπέρ, εκεί όμως δεν υπήρχε ε, στο Συμβούλιο πλειοψηφία για το κείμενο. Τις επόμενες εβδομάδες η... έγιναν συναντήσει με τις χώρες μέλη και μας προκειμένου να σταματήσει πια αυτή η μειοψηφία που μπλόκαρε τη συμφωνία. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε πλειοψηφία από το Συμβούλιο για ένα νέο κείμενο, το οποίο όμως τροποποιούσε σημαντικά διάφορα στατιστικά κριτήρια όσον αφορά τα νούμερα ε, σε σχέση με αυτά που είχαμε αποφασίσει στην αρχή. Η εφαρμογή του κανονισμού θα καθιστρούσε άλλον ένα χρόνο. Και αντί να μπορούν οι χώρες μέλη να μπορέσουν να στήσουν εξαίρεση για δύο χρόνια, παρατάθηκε αυτό για τρία συν. Η νέα πρόταση υποβλήθηκε στους σκιώδεις συζητητές για σχόλια και παρόλο που υπήρξαν επιφυλάξει, κυρίως όσον αφορά τις αλλαγέ στατιστικών σε διάφορα πιλωτικά προγράμματα, αποφάσισαν οι σκιώδεις συζητητέ ότι το νέο κείμενο θα μπορούσε να, να είναι η βάση για νέες συνομιλίε το Κοινοβούλιο προσπάθησε να είναι επικοδομητικό και να καταλήξει σε διαπραγματευτική θέση. Παρ' όλα αυτά, τι παραμονέ του τριμερού διαλόγου ενημερώθηκε το Κοινοβούλιο ότι και πάλι η Κορεπέρ δεν κατάφερε να πετύχει ειδική πλειοψηφία για το αναθεωρημένο κείμενο. Η Ισπανία, για παράδειγμα, άλλαξε τη θέση της ξαφνικά και αντί να είναι υπέρ της θέσης ήταν κατά από την ενημέρωση που έχουμε. Αυτή η ε, μειοψηφία που μπλοκάρει τα θέματα που είναι Δανία, Σλοβακία, Ισπανία και άλλες χώρες έχει σαν αποτέλεσμα οι χώρες αυτές που κανονικά θα μπορούσαν να εφαρμόσουν κάλλιστα όλες τις τροποποίησεις που προβλέπονται να μην θέλουν να το κάνουν. Αποφάσισαν να στερήσουν από τους Ευρωπαίους πολίτες από σημαντικά στατιστικά δεδομένα σε έναν από τους πιο σημαντικούς ε, τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να εξηγήσουν καν γιατί. Η κυρία Βίλστρομ θέλει να υπογραμμίσει ότι αυτή την έλλειψη επικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι κάτι απαράδεκτο. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί κάθε φορά να είναι επικοδομητικό και ρεαλιστικό. Παρ' όλα αυτά, οι χώρε μέλη στο Συμβούλιο δρούν ε, ανεύθυνα χωρίς πραγματικά να θέλουν να συνεργαστούν καλή την πίστη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Θα μπει στην ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την επόμενη εβδομάδα για να ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει τη έκθεση που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Λίμπε πριν από τι διαπραγματεύσει σε τριμερή διάλογο. Η συγκίτρια συστήνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην μπει σε ε, επόμενους τριμμένους διαλόγους με το Συμβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση αφού το Συμβούλιο δεν συνεργάζεται καλή την με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λέει η κυρία Βίλστρομ. Τώρα μια δικιά μου προσωπική παρατήρηση. Όλα αυτά δείχνουν το ίδιο και το ίδιο μοντέλο. Ότι το Συμβούλιο δεν λειτουργεί και υπάρχουν πάρα πολλοί φάκελοι για τους οποίους έχουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά. Αυτό είναι κάτι που μετά τις ευρωεκλογέ πρέπει να τακτοποιηθεί, γιατί εμποδίζει τη λειτουργία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κυρία Ντεβέλτ. Ευχαριστώ που το είπατε. Και εγώ το σκέφτηκα. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε για το Συμβούλιο. Αλλά θέλω να είμαι ευγενή. Είναι απόλυτα δυσλειτουργική εκεί πέρα. Αντικαθιστούσα την κυρία Βίξτρομ. Έχω ενδελεχή γνώση του φακέλου και είναι κρίμα. Αλλά είναι ένα είδος προσέγγισης που ισχύει. Δεν έχουμε εδώ την Προεδρία για να τις μιλήσουμε. Δεν είναι από, τους, από τα πιο μάχα θέματα, αλλά σε κάνει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Ήταν θετική η συνεισφορά σε ευαίσθητη συζήτηση όπου χρειαζόμαστε ε, αντικειμενικές προσεγγίσεις. Δεν χρειαζόταν να τσακωθούν πάνω σε αυτό. Σωστά κινήθηκε το Κοινοβούλιο. Θα το διαβιβάσουμε αυτό στην κυρία Βίξτρομ θα την ευχαριστήσουμε για τη δουλειά που έκανε και ευχαριστώ Σοφή που την αντικατέστησες. Τα σχέδιά σου έχουν Συγγνώμη, τα σχόλιά σου έχουν καταχωρηθεί. Θα ληφθούν υπόψη από το επόμενο κοινοβούλιο. Σημείο 10. Ανακοίνωση περί ενισχύσεως του κράτους δικαίου Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μιλήσει για τα βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης. Ο κ. Σλίθ νομίζω, Διευθυντής για θέματα της Ένωσης για τους πολίτες, μετανάστευση και ο κ. Κράμπιτ, Διευθυντής για τη Μονάδα Θεμελιών Δικαιωμάτων και Κράτους Δικαίου, την DG Just. Θα καταφθάσουν εδώ να καθίσουν μαζί μας. colleagues, you'll have to... Συνάδελφοι, έχετε όλη την ανακοίνωση. Χωρίς να χρονοτριβήσω, θα ζητήσω από τον κύριο Σλίθ να κάνει την πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που έχω δυνατότητα να κάνω μια μικρή παρουσίαση στην Επιτροπή σας πάνω σε αυτό το θέμα, σε αυτή την ανακοίνωση ο υπότιτλος της ανακοίνωσης είναι η κατάσταση και ενδεχόμενα νέα βήματα. Θα αναφερθώ στην κατάσταση, την τωρινή, και ο Εμμανουέλ θα αναφερθεί περισσότερο στο μέλλον. Τι θα πρέπει να διερευνήσουμε ως ενδεχόμενο στο μέλλον. Συνοψίζοντας κάπως τη γενική εικόνα που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται γιατί το κράτος δικαίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτίστως είναι θέμα αξιών. Προβλέπεται στο άρθρο 2 της συνθήκης, αναφέρεται ρητά. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι βασική αξία της ενώσεως. Υπάρχει κι άλλος πρακτικός λόγος που σχετίζεται με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και την εμπιστοσύνη που απαιτείται για αμοιβαία αναγνώριση εθνικών αποφάσεων και για την εσωτερική αγορά, άλλως ιδιαίτερο σημαντικό αυτό. Μετά υπάρχει οικονομικό στοιχείο που εμπεριέχεται στο κράτος δικαίου και προβλήματα όσον αφορά το κράτος δικαίου έχουν άμεσο κόστος και οικονομικές συνέπειες. Όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θεωρεί ότι αποτελούν μεγαλύτερη προτεραιότητα την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του του 2016 έδωσε ένα σαφές παράδειγμα για την όλη κατάσταση και προσέγγιση. Συνοψίζει η ανακοίνωση την εργαλειοθήκη όσον αφορά το κράτος δικαίου, έτσι αποκαλείται. Δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός. Τα τελευταία χρόνια είχαμε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τα διάφορα διαθέσιμα μέσα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάποια μέσα είναι οριζόντια. Τα πλέον εμβληματικά το άρθρο, είναι το άρθρο 7 από τα πιο εμβληματικά. Και τώρα έχει εφαρμοστεί όσον αφορά την Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά την Ουγγαρία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχουμε και το πλαίσιο του κράτου δικαίου που θεσπίστηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη συστηματικών απειλών όσον αφορά το κράτο δικαίου. Εν αυτή τη ενία θέλουμε να αποφύγουμε την χρήση του άρθρου 7. Να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο. Εκεί έχουμε συγκεκριμένο παράδειγμα ε, την Πολωνία που, στην οποία κοινοποιήθηκε αυτή η θέση το 2016. Ε, Μετά έχουμε τις παραβάσεις όταν υπάρχει σαφής παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εδώ έχουμε σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την ομολογία του δικαστηρίου και θα έχουμε και συνέχεια σήμερα. Εκεί αναγνωρίζει τη σημασία του κράτους δικαίου για την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βασικό κομβικό στοιχείο του όλου ζητήματος που συζητούμε. Η εργαλειοθήκη συμπεριλαμβάνει και τομιακά μέσα που σχετίζεται με τα κράτη-μέλη. Έχουμε το μηχανισμό κοινοποίηση που ακόμα εφίσταται σε δύο κράτη-μέλη. Πρέπει να δούμε και τομιακά τι γίνεται όσον αφορά τις πολιτικές και εκεί έχουμε πρόταση στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου που θεσπίζει μηχανισμό όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από πλευράς παραβάσεων του κράτους δικαίου για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχουν και εργαλεία με περισσότερο γενική προσέγγιση που αφορούν το κάτω δικαίου, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είναι προφανές παράδειγμα. και το σύστημα βαθμολόγησης για τη δικαιοσύνη που άπτεται του κράτους δικαίου και έχουμε και άλλα εργαλεία και μέσα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει και τα χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να παγιώσουν το κράτος δικαίου και τις συναφείς υποδομές, τα διεθνωτικά ταμεία και υπηρεσία στήριξης των διαστατικών μεταρρυθμίσεων. Και υπάρχει και το θέμα της γειτονίας. Εκεί το κράτος δικαίου στις διαπραγματεύσεις είναι πολύ σημαντικό και κυρίως στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα και αρχές που διαφαίνονται. όσον αφορά τη μελλοντική μας προσέγγιση. Καταρχάς, έχει νομικό συμφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το τομέα και τα άλλα κράτη-μέλη για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου. Μετά υπάρχει μεγάλη ευθύνη των κρατών μελών αυτών καθεαυτών και η πρώτη προσφυγή θα πρέπει να γίνεται μέσω εθνικών μέσων για την επίλυση ζητημάτων, να μην γίνεται αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών. και πρέπει να υπάρχει αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη που θα εφαρμόζεται. Τέλος, στόχος, ο στόχος δεν πρέπει να θεωρείται που δεν είναι ότι έχει μορφή κυρώσεων, αλλά είναι προσπάθεια επιλύσεως πραγματικών προβλημάτων. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ε, συγκεκριμένους πρακτικούς στόχους και λειτουργίες, συνοψίζοντας την όλη κατάσταση. Να σας πω λοιπόν ότι καταρχάς Έχουμε εξελίξιμη ανάγνωση του τι σημαίνει το κράτος δικαίου. Μετά έχουμε ένα οικοσύστημα ε, του κράτους δικαίου που έχει ε, εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια με γρήγορους ρυθμούς. Και τέλος, εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε βελτιώσεις όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου και πώς εξασφαλίζεται αυτή η εφαρμογή. Έχουμε ακόμα δουλειά. Ο Εμμάνουελ θα πει κάποια πράγματα όσον αφορά τις ε, διεξόδους, τις μελλοντικέ που έχουμε εντοπίσει. Σας ευχαριστώ πράγματι για να διευκολύνουμε την διαδικασία αυτή. Έχουμε τονίσει κάποιες πιθανές ε, διόδους ε, και αυτές διαχωρίζονται σε τρεις τύπους, τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την προαγωγή το θέμα είναι δηλαδή πως θα προωθήσουμε μια κουλτούρα κράτους δικαίου και συγκεκριμένα πως θα προωθήσουμε την καλύτερη γνώση των ε, υφιστάμενων ευρωπαϊκών διατάξεων που αφορούν το κράτος δικαίου. Ένα από τα μαθήματα που μάθαμε από το παρελθόν είναι ότι οι υφιστάμενες διατάξεις ε, δεν είναι πολύ γνωστές σε εθνικό επίπεδο και όχι μόνο αυτό, αλλά και ε, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις έρευνες της Επιτροπής της Βενετίας ε, και άλλων. Βασική πρόκληση είναι το πώς ακριβώς θα προωθηθούν αυτές οι προδιαγραφές στο εθνικό επίπεδο. Τα εθνικά κοινοβούλια ειδικά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Ο ρόλος επίσης του διακοινοβουλευτικού διαλόγου ήταν Ε, βασικό κομμάτι της δουλειάς που γίνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Επίσης ε, πρέπει στο πλαίσιο αυτό να δούμε το θέμα της ε, αναθεώρησης από τους ομοτήμους που προτείνεται από κάποια κράτη-μέλη. Επίσης το θέμα της, των ανταλλαγών μεταξύ δικαστών, ε, δικηγόρων, ε, της κοινωνίας των πολιτών για να προωθηθούν ε, καλύτερα αυτά τα θέματα για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτές τις πηγές πληροφοριών και βεβαίως σημαντικό θέμα είναι η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να εντείνουμε αυτήν την ε, συνεργασία. Τέλος, μία άλλη πρόκληση που δεν πρέπει να υποτιμούμε είναι πώς θα επικοινωνούμε καλύτερα με το κοινό. Θυμάμαι ότι είχε οργανώσει η Επιτροπή σας ένα σεμινάριο με τον Διεθνή Δικηγορικό Σύλλογο που είχαν παρουσιάσει κάποια μικρά κλιπ επίσης για το κράτος δικαίου, κάτι σημαντικό για να εξηγηθεί στο κοινό. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους δικηγόρους, αλλά αφορά τους πάντες. Ο δεύτερος πυλώνας ε, αφορά την πρόληψη. Πρέπει να βελτιώσουμε ε, την ε, γρηγορότερη ανείχνευση προβλημάτων, έγκαιρη ανείχνευση για να αποφευθεί η κλιμάκωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη τα οποία προβαίνουν σε μεταρρυθμίσεις συνταγματικές ή κατά τις μεταρρυθμίσεις θα συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές αυτές προδιαγραφές και βασική πρόκληση εδώ πέρα είναι το πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια πιο βαθιά γνώση αναχώρα και συγκριτική ε, των ε, κρατών μελών. Η ανακοίνωση μας ζητάει ακριβώς ε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο διάλογο με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα βαθμολογίας ή το ευρωπαϊκό εξάμεινο περαιτέρω για να περιλάβουμε ζητήματα κράτους δικαίου. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις βεβαίως και ιδέες μεταξύ των οποίων το σύμφωνο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένας άλλος ε, τομέας ε, όσον αφορά την πρόληψη είναι το πώς θα υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία κάνουν μεταρρυθμίσεις ε, μέσω τεχνικής αρρωγής. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα κράτη-μέλη έχουν πολλά να μάθουν το ένα από το άλλο, παραδείγματος μέσω της ε, υπηρεσίας στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, Παραδείγματο χάρη ναι, η Κομισιόν χαρτογραφεί το δικαστικό τοπίο που υπάρχει σε πόλεις, περιφέρειες κτλ. Ε, με το να φέρνει μαζί ειδικού από τα διάφορα κράτη-μέλη που κάνουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Ο τρίτος πυλώνας για την πιθανή μελλοντική δράση είναι η ε, δυνατότητα αντίδρασης, η δυνατότητα να υπάρξει δηλαδή μια αποτελεσματική αντίδραση όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό ε, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους εθνικούς ε, μηχανισμούς όπως έχουμε τονίσει, έχει τονίσει και ο πρώτος αντιπρόεδρος το βασικό εδώ πέρα είναι να βελτιώσουμε τη δυνατότητα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις που απαιτούν διάφορες απαντήσεις και τα εργαλεία που απάντησε, που ε, ανέφερε η Κομισιόν παρέχουν μια δυνατότητα ευρύτατων αντιδράσεων. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες εδώ πέρα. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν μας ζητάει να σκεφτούμε το πώς ακριβώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό και πώς ε, θα υπάρξει μια διάδοση σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει και η πρόταση της ε, Κομισιόν για την προστασία των οικονομικών σφαίρων της κοινότητας από την έλλειψη ε, κράτους ε, δικαίου και βεβαίως η ανακοίνωση προτείνει να σκεφτούμε το τι γίνεται στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διάλογος που βασίζεται σε λεπτομερείς αναλύσεις και θα μπορούσαμε να δούμε αν απαιτούνται κάποιες άλλες ρυθμίσεις για το πλαίσιο αυτό, να δούμε παραδείγματος χάρη πώς θα ενταθεί η πληροφόρηση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Καναλίγοντας λοιπόν, ε, είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα η δική σας Επιτροπή νομίζω ότι είναι σαφές πως ε, το κράτος δικαίου είναι εκείνη η ευθύνη ε, όλων των κοινωτικών οργάνων και πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σίγουρα θα συνεχιστεί η συζήτηση από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά για τους μαχητές υπέρ του κράτους δικαίου Επιτρέψτε μου να σας πω έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ πάντως. Πραγματικά. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς προχωράει η μεταρρύθμιση και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς τα πράγματα. Να το ξέρουν και αυτοί που δεν θα επανέλθουν. Σόφι, πώς τα βλέπεις εσύ αυτά που άκουσες και η Τζούντιθ μετά. Ευχαριστώ Κλοντ. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κράβιτ και τον κύριο Σλίθ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ό,τι θα πω δεν το λέω σε εσά προσωπικά. Έτσι, καταλάβατε τι σας περιμένει. Να είσαι ευγενής, λέει ο πρόεδρος. Ξέρω για πολλά χρόνια τι προσπάθειες έχετε κάνει για αυτό το θέμα, οπότε δεν έχω να επικρίνω σας προσωπικά. Αλλά το θέμα είναι, μια που μιλάμε για μαχητές, σας μιλήσουμε καλύτερα για μονομάχους. Πού είναι ο κύριος Τίμερμαντς? Έτσι θα προστατεύσει το κράτος δικαίου. Μα είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία αυτή. Πούντος. Και γιατί παρουσιάσετε αυτό το θέμα την πρώτη τελευταία εβδομάδα εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα θα έρθουν τον Ιούνιο όταν ε, θα διαμορφώνεται το νέο Κοινοβούλιο. Έτσι θα χειρίζεται αυτά τα θέματα ο κύριος Τίμερμαντς. Και εδώ δεν μιλάω και μόνο για τον κύριο Τίμερμαντς, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπεύθυνο για το κράτος δικαίου, μιλάω και για τον κύριο Τίμερμαντς που είναι υποψήφιος για πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κακή στιγμή αυτή η συγκυρία. Έπειτα, ξέρω, στον τίτλο, παρόλο που άκουσα τον κύριο Κράμπιτ να μιλάει για ολόκληρο το φάσμα του άρθρου 2, δεν είναι στον τίτλο. Ο τίτλος μιλάει μόνο για το κράτος δικαίου και επικεντρώνεται στα όργανα, δικαστική εξουσία κλπ. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείναμε ολόκληρο το DRF δηλαδή δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα, όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 2. Οπότε, τι προσθέτει. Μα συνοψίζει ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ωραία, το είχαμε αυτό. Και μετά ζητάει συνεισφορά. Προσπάθησα να καταλάβω πού μπορεί ο κόσμος να στείλει ό,τι θέλει. Έχω εδώ αντίγραφο για την συμφωνία αυτή από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας το δώσω. Μπορείτε ίσως να το στείλετε στον κύριο Τίμερμανς. Γιατί πολλά από αυτά που αναφέρατε κι εσείς στην παρουσίασή σας υπάρχουν στην πρόταση. Και ο κύριος Τίμερμανς τότε, όταν εμείς ψηφίσαμε, είπε δεν το χρειαζόμαστε γιατί έχουμε την εργαλειοθήκη που χρειαζόμαστε. Ε, λοιπόν, όχι. Τρία χρόνια μετά, Πολωνία, Ουγγαρία, άλλες χώρες, Μάλτα, Σλοβακία, Ρουμανία, ό,τι θέλετε. Και βλέπω ότι παρά την ανακοίνωση αυτή που έχουμε μπροστά μας τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εργαλειοθήκη της έχει το άρθρο 7, αλλά αρνήθηκε, ό,τι απέτυχε να τον αργοποιήσει, αρνήθηκε να τον αργοποιήσει για την Ουγγαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε τρεμερείς διαλόγους για αξίες, διάλογο κτλ. Και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μειώσει τις ε, κυρώσεις όταν δεν εφαρμόζονται αυτά που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έπειτα η αιρεσιμότητα, από ό,τι βλέπω, επίσης κατεβάζει το επίπεδο όσον αφορά το κράτος δικαίου σε μια καθαρά τεχνοκρατική άσκηση, ενώ πρόκειται για πολιτική. Και δεν εννοώ πολιτικά αντική, ενώ πολιτική ευθύνη, είναι πολιτική προτεραιότητα. Ο κύριος Τίμερμανς θα έπρεπε έγκαιρα πέρυσι να έρθει και να μας τα παρουσιάσει στην Ολομέλεια ή έστω εδώ, στη Λίμπε. Και όχι μια εβδομάδα πριν τελειώσουν οι εργασίες μας. Δεν ξέρω, θα κάνει προεκλογική εκστρατεία μάλλον ο κύριος Τίμερμαν τώρα, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Λοιπόν, αν αυτά έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μην μας εκπλήσει που ουσιαστικά όλη αυτή την ιστορία την αναθέτουμε στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε δημοσιονομικές αρχές και δεν ξέρω που αλλού, ενώ θα έπρεπε να είχαμε έναν ισχυρό μηχανισμό που να καλύπτει όλες τις χώρες μέλη, που να είναι ενεργός αυτός ο μηχανισμός συνέχεια. Συνεπώς, αν μη τι άλλο, από πλευράς χρονοδιαγράμματος θα ζητούσα έντονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καταλήξει συμπεράσματα τον Ιούνιο. Είναι εμβληματικό θέμα, έτσι να το δείτε κι εσείς. Και παρουσιάστε το μετά την 1η Νοεμβρίου με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα θέματα αυτά τη δημοκρατία του κράτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μην το κατεβάσετε σε επίπεδο ενό τεχνοκρατικού εγχειρήματο, να το διατηρήσετε σε επίπεδο εμβληματική πολιτική και να το αφήσετε και την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρον αυτό το πώ θα το παρουσιάσει το Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο θα είναι εκεί. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Θα δούμε ποια είναι η άποψη των συναδέλφων. Η Τζούντιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα το Συμβούλιο ξανά μίλησε για την Ουγγαρία, για την Πολωνία. Ξανά δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα και το τι πρέπει να γίνει. Την περασμένη εβδομάδα επίσης συμπεράναμε, ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβούλιο μάλλον λέγαμε ότι οι διαπραγματεύσει για το δημόσιο ε, εισαγγελέα δεν πηγαίνουν πουθενά. Και ε, τελικά στο Συμβούλιο ε, παραμελούν εντελώς το Κοινοβούλιο. Ε, μην δεχόμενοι έναν υποψήφιο. Έχουμε θέματα κάτω δικαίου. Ξέρω ότι μιλάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφερόμενη στο Συμβούλιο, τέλος πάντων. Το ξέρω αυτό. Αυτή η ανακοίνωση δεν δείχνει ότι είναι επίγον το θέμα, παρόλο που είναι επίγον το θέμα και θα ήταν μια πανεύκολη λύση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείξει ότι είναι το θέμα. Πρέπει να ξεκινήσει η πραγματική συζήτηση με το Κοινοβούλιο μετά την έκθεση της κυρίας Ινφελτ για το πακέτο DRF. Έπρεπε να γίνει αυτό. Ήταν πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου, έκθεση νομοθετικού περιεχομένου. Και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι τελικά ε, κάτι που προσπαθεί να χρονοτριβήσει. Δηλαδή να περάσουν οι ευρωεκλογέ και να μπούμε σε διαφορετικό πολιτικό χώρο. Και αυτό είναι προβληματικό. Διότι αυτό κάνει και το Συμβούλιο με τους Ούγκρους και τους Πολωνούς που κολλησιεργούν να κερδίσουν χρόνο, να μην γίνει συζήτηση πραγματική στο Συμβούλιο μέχρι μετά τις εκλογές και οι Ρουμάνοι μπλόκουν την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία ε, Εισαγγελία. Και τώρα μα δίνει μια ανακοίνωση καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θέλουμε να υπάρξει εφησυχασμό. χρειαζόμαστε δράση. Πρέπει να δώσουμε στου Ευρωπαίου πολίτε που πάνε να ψηφίσουν σε κάνα δύο εβδομάδε, ότι αυτό είναι ένα θέμα το παίρνουν στα σοβαρά. Αυτό που είπε η κυρία Ιντφέλτ ότι αυτό δεν είναι προσωπικό ισχύει και για μένα. Αυτά που λέω δεν είναι προσωπικά απευθυνόμενα σε εσά, αλλά έχω απογοητευτεί πραγματικά πολύ διότι δεν φαίνεται εδώ η ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε τάχιστα. είναι πήγον το θέμα. Το Κοινοβούλιο προσπάθησε να σας πλησιάσει και ξεκάθαρα είπε στο Συμβούλιο ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μόνη της που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και οι τρεις έχουμε αυτή τη θέση. Αλλά θέλω εσείς να είσαστε θεματοφύλακα της συνθήκες και κάθε φορά που προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις όσον αφορά το δικαστικό σύστημα χάνουμε διότι απομακρυνόμαστε από την πολιτική απόφαση. Τέλος, Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια υπέροχη ανακοίνωση το 2003 με τίτλο «Σεβασμός και προώθηση των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση». Και σε αυτή την ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι το άθρο 7 είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή ανάλυση των συνθήκων. Είναι αυτό που αφορά τα πάντα που συμβαίνουν ένα κάτω μέλο. Θα ήταν καλό αν η ανακοίνωσή σα αυτό το ελάμβανε υπόψη και να κάνατε συγκεκριμένες προτάσεις, διότι θα το λύσουμε αυτό μέσω συνενέσεις. Είδαμε χτες ότι οι Ολλανδικές μυστικές υπηρεσίες δεν θέλουν να συνεργαστούν πλέον με τις Αυστριακές μυστικές υπηρεσίες, διότι είναι ένα τμήμα της αυστριακής κυβερνήσεως πολύ κοντά στου Ρώσου. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα κράτους δικαίου και πρόβλημα ασφαλεία και θα πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τονίσω κι εγώ ότι δύο φορές το Κοινοβούλιο έχει παραμεριστεί και για το Άθρεπτα και την Ουγγαρία έπρεπε βάσει των προνομίων να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να παριστάμεθε. Για τα προνόμια, βάσει των προνομίων που έχουμε, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προνόμια. Είναι σημαντικό. Τι λέει για τις παρούσες εξουσίες όταν αναλύεται μελλοντικέ εξουσίες. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Χουάν, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κλοντ, ευχαριστώ και εσάς που στο τέλος εδώ, προς το τέλος της θητείας, θέσατε τον υπαριθμό ένα θέμα, για να το πω ομά, το κράτος δικαίου. Μας νοιάζει, πάντα μας ένοιαζε, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχαμε λόγο γι' αυτό. Είχαμε πολλές οπισθοχώρησεις και καταστάσεις. πέδουξαν επιδείνωση όσον αφορά το δικαίου και τη βούληση συμμόρφωση σε αρκετά κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο λοιπόν είναι δυσλειτουργικό όσον αφορά τις λήψεις αποφάσεων. Και όλο και περισσότερο αμελεί το θέμα αυτό, το κάτω δικαίου. Και βάσει των όνων αυτών που είπαμε, και αυτά που τονίστηκαν του συναδέλφου, να πω και εγώ ότι στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε την πολιτική βούληση για να υπάρχει συμμόρφωση με τον νόμο από πλευρά κρατών κυβερνήσεων. Κατών μελών και κυβερνήσεων των κατών μελών. Που όλο και περισσότερο παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχουν ε, διαδικασίες επί παραβάση και αρκετές. Υπάρχει και το ΔΕΚ. Αρκεί κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, υπήρχε ο φόβος του Θεού. Όχι πλέον. Κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, τα κράτη-μέλη είχαν και εδώ δεν ήθελα να δακτυλοδεικτούν, να τους δακτυλοδείχνουν ότι παραμελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όχι πια. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεκάρα δεν δίνουν υγεία διαδικασίες επί παραβάση. Ούτε καν για τις αποφάσεις του ΔΕΚ. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε το κύρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πώ θα υπάρχει πολιτική βούληση συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Στην προηγούμενη θητεία του Ευρωκοινοβουλίου εκτενώς συζητήσαμε το άθρο 6 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως που καθορίζει την εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όχι πλέον. Έχει βγει από την εικόνα αυτό. Με αυτό τι τρέχει. Υπήρχε και διάλογος μεταξύ ευρωπαϊκών ενόμων τάξεων για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπήρχε εικόνα διαλόγου μεταξύ ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του ΔΕΚ στο Λουξεμβούργο και συζητήσεις με τα δικαστήρια και τα συνταγματικά δικαστήρια των κρατών μελών. Ε, φαινόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας παράγων, ένα μέλος επρόκειτο να γίνει μέλος του, του συστήματος της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή είναι η εντολή που δίνει το άρθρο 6. Και βέβαια είχαμε και γνωμοδότηση του ΔΕΚ που θέτει τις προδιαγραφές και τα πρότυπα. Θεώρησε το ΔΕΚ ότι δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε χωρίς τροποποίηση τη συμφωνίας που συνήφθη από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθέτησε. Δίγησε το μονοπάτι για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έκτοτε όμω, δεν το κουβεντιάσαμε. Έσβησε από την εικόνα το θέμα. Δεν το κουβεντιάζουμε καν. Μα τι θα γίνει. Τι πρόκειται να γίνει ούτω ώστε να πετύχουμε το στόχο του άρθρου 6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Πήρκετε. Δεν θέλετε το λόγο. Ε, δεν σκόπευα, αλλά τώρα θέλω να προσθέσω κάτι. Λίγο πολύ σαφέστατα υπόθηκε. Το κύριο πρόβλημα το οποίο βλέπουμε δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που θα ήθελα πιο πολιτική, πολιτική ανάμιξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο, είναι οι χώρες μέλη. Μεμονωμένη καθεμία, αλλά και το Συμβούλιο ολόκληρο ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν καταφέρει να αναβάλει τις ευθύνες του για το τι συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε και στην επόμενη θητεία πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να ελέγξουμε κάπως καλύτερα αυτά που συμβαίνουν στο Συμβούλιο, να μάθουμε περισσότερα για τις διαδικασίες που ακολουθούν, γιατί τελικά εκείνοι είναι που μπλοκάρουν τα πάντα. Και αυτό επιπλέον μετά όσα είπαν οι συνάδελφοι. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν στην επόμενη θητεία. Τι κάνει το Συμβούλιο, τι σόι θεσμικό όργανο είναι. Και είναι τελικά ακόμα ένα ευρωπαϊκό όργανο ή μήπως πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Παίρνω το λόγο γιατί δεν συμφωνώ για το κράτος δικαίου και αυτά που είπε ο Κλοντ και άλλοι. Εμείς ελέγχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε όσον αφορά το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους άλλους. Η δημοκρατία τι είναι. Είναι πρώτα απ' όλα ο έλεγχος της εξουσίας και όχι ο έλεγχος μέσω της εξουσίας. Τώρα, για την πολιτική αποσία του κύριου Τίμερμαντς τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Στην Κυριακή ήταν στη Βαρσοβία ε, για την εκστρατεία του νέου κόμματο που ονομάζεται Άνοιξη και βρίσκεται αριστερά της αριστεράς στην Πολωνία και είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Χρησιμοποιεί ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για να προωθήσει τη δικιά του πολιτική θέση στην προεκλογική εκστρατεία που είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών ο Spitzenkandidat. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να εκφράσουμε την ανησυχία μας ότι δεν κάνει αρκετά ο κύριος Τίμερμανς, ότι δεν είναι δραστήριος σε αυτή την εποχή. Τώρα όσον αφορά το δικό μας έλεγχο της εξουσίας, πρέπει να σεβόμαστε τη συνθήκη. Γιατί, Γιατί αυτό που ρώτησε ο Χουάν Φερνάντο, ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να εκτελούμε την πολιτική μας βούληση αντιφάσκει με το πνεύμα του κράτους δικαίου. Γιατί εμείς πρέπει να δρούμε στα όρια που μας βάζει ο νόμος, η συνθήκη δηλαδή. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αν το άρθρο 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι μόνο σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις μπορούμε να δηλώσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία σε μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς για να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός στην ποικιλομορφία των νομικών μας συστημάτων. Οπότε, με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση ε, για το κράτος δικαίου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ευθανασία, για παράδειγμα, που επιβάλλεται μερικές φορές στις κατοχώρες ή σε άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό μέλλον και πρέπει να σεβόμαστε ένας τον άλλον. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για εσάς. Εσείς γελάτε. Καλά, αλλά για μένα ή σε άλλες χώρες. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα κοινό μέλλον και πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για σας. Για εσείς γελάτε. Καλά, αλλά για μένα η θανάτωση ανθρώπων ο σύντροφός τους, τους θανατώνει ας πούμε σε μια κλινική όταν αυτή η ευθανασία επιβάλλεται. Για μένα η ζωή είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Αλλά εντάξει, εσείς έχετε διαφορετικές θέσεις. Ωραία. Αν είμαστε μια κοινότητα, τότε πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλον και να σεβόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Γιατί η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ο έλεγχος των χωρών, είναι η αλληλεγγύη, είναι η βοήθεια προς τις χώρες. Ελπίζω λοιπόν ότι η αποστολή μας για έλεγχο του κράτους δικαίου στην επόμενη θητεία θα γίνει με αυτοέλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελέγχοντας τα θεσμικά όργανα και όχι να ελέγχουμε τις δημοκρατικές αποφάσεις που λαμβάνονται στις διάφορες ε, χώρες από τους πολίτες. Σας ευχαριστώ βεβαίως. Ε, ρώτησα τη γραμματεία αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελευταίο θέμα για την πολιτική άμυνα ή κάτι πιο ήπιο εν πάση περιπτώσει. Αλλά όχι, μου είπαν. Λοιπόν, πάμε. Φουλ κράτος δικαίου και ας τα αφήσουμε για την επόμενη θητεία θυμίζουν εδώ πέρα τη συνεδριάση για Ουγγαρία, Πολωνία και τα σχετικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά είναι αυτά έτσι, ωραία. Περνάμε τώρα ξανά στους συναδέλφους μας για μία απάντηση. Έτσι είδατε πώς είναι η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάποια θέματα. Βεβαίως ε, το κείμενο της ανακοίνωσης ε, προφανώς ε, αυτή τη στιγμή είναι εντάξει ένα έγγραφο και έτσι φαίνεται ότι έχουν τα πράγματα και προφανώς αναμένουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες ιδέες αλλά ακόμα και έτσι ναι, δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα τελειώσουν. Με πιο συγκεκριμένες ιδέες προς ε, συζήτηση. Το στυλ αυτό της ανακοίνωσης βεβαίω. Λοιπόν, για την επόμενη επιτροπή τώρα αν ανησυχούν εδώ πέρα οι, μαχητές ε, του κράτους ε, δικαίου. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά μας εμάς να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά ελπίζω ότι αυτό το οποίο θα προκύψει από το κείμενο είναι αυτή η αίσθηση μιας ορμής ε, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχει υπάρξει εδώ πέρα πραγματικά μια διαδικασία κατά την οποία η Κομισιόν μαθαίνει και όσον αφορά την έκταση των προκλήσεων, αλλά και το πώς ε, θα τις αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι έχουμε μάθει πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, παραδείγματος χάρη. Μιλήσαμε για αυτούς τους τρεις τίτλους, ε, θέλετε, την πρόληψη, την προώθηση και την αντίδραση. Και συνδέονται αυτά τα πράγματα και ένα από τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι ότι για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε εντόνως ε, Όσο περισσότερο έχουμε προωθήσει εκ των προτέρων μια κοινή αντίληψη, τόσο περισσότερο έχουμε λύσει τα προβλήματα εκ των προτέρων και ευκολότερη είναι και αντίδραση. Λοιπόν, νομίζω ότι τέτοια ζητήματα είναι τομείς όπου σε μια δεύτερη φάση πρέπει να ε, γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Και Νομίζω ότι θα συνεχίσει και στην επόμενη Κομισιόν αυτή η πορεία. Θα μου προξενούσε εντύπωση το αντίθετο. Ναι, για την αίσθηση αυτή της ανυπομονησίας, αν θέλετε, και του κατεπήγοντος πράγματι συμφωνούμε. Ως προς αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι mm-hmm. σημαντικό να το δούμε ως κάτι το θετικό, μια θετική ενέργεια και χάρη σε εσά. νομίζω έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο σε λίγα χρόνια θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι το πιο θετικό, θετική ενέργεια για εμάς για να έχουμε περισσότερο κράτος δικαίου. Οπότε νομίζω ότι βεβαίως θα θέλαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα, αλλά πρόκειται για μια κοινή μας ε, ευθύνη. Βλέπουμε ότι με την προσέγγιση αυτή έχουμε μια καλή μέθοδο για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι μια κοινή μας ε, ευθύνη. Όπως σημειώσατε έχουμε κάποιες προκλήσεις στο Συμβούλιο, σε κάποια κράτη-μέλη. Πρέπει όμως να δημιουργηθεί μια δυναμική, μια δυναμική οποία θα έχει κάποια αποτελέσματα και τέλος για την αίσθηση αυτή του κατεπήγοντος. Κοιτάξτε, ακριβώς έπρεπε να δράσουμε λόγω της κατεπήγουσας κατάστασης. Οπότε ξεκινήσαμε διαδικασία σε επιπαραβάση όπω όπως και στην Ουγγαρία και στην ε, Πολωνία προτείναμε έναν νέο κανονισμό για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού σε περιπτώσεις γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και να με συγχωρείτε νομίζω ότι πριν από πέντε χρόνια ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσε ε, να είναι δυνατόν να προτείνουμε κάτι τέτοιο και χάρη σε εσά, χάρη στην στήριξή σας ε, καταφέραμε να προχωρήσουμε Βεβαίω οι διαπραγματεύσει ε, συνεχίζονται, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Οπότε είναι σημαντικό όταν ε, μιλάμε για νέους μηχανισμούς να μην αποκλίνουμε από τα πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να συζητήσουμε για νέους μηχανισμούς και τα λοιπά, αλλά πρέπει να δράσουμε. Και αυτό ακριβώς προσπάθησε να κάνει η ε, Κομισιόν. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε επί τη ευκαιρία. Όταν η Κομισιόν δρά, για θέματα κράτους δικαίου είναι τελείως ε, ουδέτερη. Είναι μια απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων. Σας ευχαριστώ. Θα σας ρωτούσα αν έχετε ιδέα το τι θα κάνετε μετά τον Ιούνιο, αλλά η Σόφη θα έχει την τελευταία κουβέντα. Ορίστε Σόφη. Um, Ερώτηση. Γιατί δεν το κάνετε μια πραγματική διαβούλευση. Σε τόσο άλλα θέματα αυτό κάνατε. Γιατί δεν ανοίγεται μια πλήρη διαδικασία διαβουλεύσεων. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν. Έτσι. Το Κοινοβούλιο θα το κάνει σίγουρα με κυβερνητικές οργανώσεις, κυβερνήσεις, ακαδημαϊκοί, όλοι. Γιατί δεν ξεκινάτε μια πραγματική διαδικασία διαβουλεύσεων. Κοιτάξτε, Πρόκειται περί ανοιχτή διαδικασία, κατά κάποιο τρόπο, σε κανονικέ διαβουλεύσει που δεν υιοθετούνται όμω σε επίπεδο. Οι κανονικέ διαβουλεύσει δεν υιοθετούνται σε επίπεδο κολεγίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι κάπω υψηλότερο. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε φορείς να εκφράσουν ιδέες ευπρόσδεκτη αυτή η συνεισφορά, η κύριε Ντφέλτ. Σωστή κανονική διαβούλευση. Δεν ξέρω αν υιοθετείται από το σώμα, το κοινοβούλιο, όχι. Κάτι που ανακοινώνεται, που είναι δημόσιο, έχει χρονοδιάγραμμα, προθεσμίε, καθορισμένε ερωτήσει. Διαβούλευση, όπω έκανε επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε. Ρητορική δήλωση, λέει ο πρόεδρο αυτή. Ευχαριστώ του δύο συναδέλφου ε, για που ήρθαν εδώ να μα μιλήσουν και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους στα διάφορα δεν υπάρχουν διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση δεν υπάρχει επόμενη συνεδρίαση. Θα μπούμε στη μαύρη μα τρύπα. Είδατε τη μαύρη τρύπα χθε στην τηλεόραση. Η μαύρη τρύπα η δική μας είναι η επόμενη θητεία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα όμως. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι το τέλος εδώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.